το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, ξεκινώ ευχαριστώντας τους σκιώδεις ηγητέ όχι μόνο για την επικοδομητική συνεισφορά του, στη σύνταξη τη εκθέσεως, αλλά για πραγματική αφοσίωση και προσπάθεια για την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμηση κατά των διακρίσεων. Το 2000 ανήκα σε μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικό δίκτυο που ζητούσε την έγκριση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Όταν οι δύο οδηγίε για την ισότητα υιοθετήθηκαν, θεωρήσαμε ότι ήταν μια ιστορική στιγμή, διότι η διάκριση κατά άλλων ανθρωπίνων όντων είναι μία, μία από τι πιο αξιόμεμπτε συμπεριφορέ. 16 χρόνια μετά έχω το προνόμιο σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιολογήσω το πώς η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση έχει εφαρμοστεί. Το 2000 ε, τα κράτη-μέλη υποχρονόταν να προστατεύσουν τους ανθρώπους κατά των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής ε, κατάρτισης. Δεν εκπλήσει κανέναν ότι ναι μεν κάποια κράτη-μέλη ξεπέρασαν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας επεκτείνω την προστασία κατά των διακρίσεων και σε άλλου τομεί, όπω είναι η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε. Άλλα κράτη-μέλη πόρο απέχουν από την εφαρμογή τη οδηγία στο ελάχιστο επίπεδο. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη που υπάρχει για τη συλλογή στοιχείων περισσότητα και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να διευκολυνθεί η απόδειξη ε, τη ανισότητα και τη διάκριση, κυρίω έμεση διάκριση. Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των επιπέδων διακρίσεων που ε, αναφέρονται και εκείνων που πραγματικά σημειώνονται. Η ευαισθητοποίηση με τη βοήθεια φορέων για την ισότητα και των κοινωνικών εταίρων είναι υψίστη σημασία σε όλα τα επίπεδα, τα κοινωνικά, διότι τα ίδια τα θύματα έχουν πρόβλημα ε, για να αναγνωρίσουν τη διάκριση και πολλοί δε μάλλον να την καταπολεμήσουν. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά ε, το ρόλο που παίζουν οι φορείς την ισότητα για την ευαισθητοποίηση και συλλογή στοιχείων, τη βοήθεια που δίνουν στα θύματα αλλά και σε εργοδότε να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν την πολιτική του σύμφωνα με τι απαιτήσει περί ισότητας. Η αμεροληψία τέτοιων φορέων θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η δραστηριότητά τους να υποστηρίζεται και μέσω επαρκούς χρηματοδοτήσεως. Θα ήθελα ιδιαίτερως να τονίσω το θέμα της πολλαπλής διάκρισης που πολύ συχνά είναι μια συνέπεια της ύπαρξης κατακαιρματισμένων προτύπων και κανόνων στα κράτη-μέλη. Εάν για ένα είδος της διακρίσεως είναι δύσκολο τα θύματα να κατανοήσουν ότι είναι θύματα και να δράσουν, μπορούμε να φανταστούμε τη δυσκολία έχουν όταν αντιμετωπίζουν πολλαπλές ε, διακρίσεις. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ακόμα περιορισμένη σε πολλές περιπτώσεις διακρίσεων και η έκθεση συστήνει ένθερμα στα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τα θύματα μπορούν να έχουν ε, νομική αρρωγή και συμβουλές σε όλες τις φάσεις της ένομης αυτής της νόμης διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης και της εμπιστευτικής βοήθειας και παροχή συμβουλών από τους αρμόδιους φορείς. Και η νομική αποκατάσταση δεν είναι μόνο σημαντική για τα θύματα, αλλά έχει και εκπαιδευτικό αντίκτυπο επί της κοινωνίας, διότι η εκδίκαση υποθέσεων και επαρκή εκπροσώπηση των θυμάτων εξακολουθεί να είναι προβληματική σε κάποιες περιπτώσεις και ζητούμε τα κράτη-μέρη να βρουν τρόπους να βοηθήσουν τα θύματα, όπως μέσω εξαιρέσεων, μειώσεων από φορολόγηση, νομικής αρρωγής και βοήθειας από ειδικευμένους ΜΚΟ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η νομική θέση των ΜΚΟ με νόμιμα συμφέροντα σε διάφορες ε, δικαιοδοσίε. Θα πρέπει να γίνονται αλλαγή βελτίστων πρακτικών των κρατών μελών. Είναι προαπαιτούμενο. Πρέπει να δεχτούμε ότι η καταπολέμηση κάθε μορφή διάκριση πρέπει να γίνει αποδεκτή, παραδεκτή και να υποστηρίσει το Κοινοβούλιο μεγάλη πλειοψηφία αυτή την έκθεση. Σα ευχαριστώ. Κυρία Βέμπερ, το λόγο εξ Επιτροπή έχει η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Βέμπερ, την εισηγήτρια, που εκπώνησε αυτή την περιεκτική αξιολόγηση της εφαρμογής ε, της ε, οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση. Διάκριση όπου και αν οφείλεται, δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι οι οδηγίε κατά των διακρίσεων εφαρμόζονται αποτελεσματικά στα κράτη-μέλη, προκειμένου να προωθηθεί μια δικαιότερη, πιο χωρί αποκλεισμού κοινωνία, με δυνατότητε στην αγορά εργασία για όλου του συμπολίτε και προβλέπεται και στα, στο κοινωνικών δικαιωμάτων ότι θα πρέπει να διευρυθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασία και να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση σε όλου του κλάδου και με την καλύτερη ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση των φαινομένων διακριτική μεταχείριση. Είναι αναφυσβήτητο ότι πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δημιουργούν προβληματισμό και ανησυχίε. Με βάση το Ευρωβαρόμετρο του 2015 για τι διακρίσει, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ευρία αντίληψη φαινομένων διάκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 64% όσο όσων έδωσαν απαντήσεις εξέφρασαν ανησυχίες για διακρίσεις λόγω εθελοντικής καταγωγής, 56% ε, λόγω γενετήσεων προσανατολισμού ε, και λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και κάποια πρόοδο. Ε, το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι πολίτες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τα δικαιώματά τους στον τομέα αυτό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα για να βελτιωθεί η εφαρμογή της ισότητας. Και μάλιστα μετά την ε, έκθεση εφαρμογής ε, του 2015 για την εφαρμογή της οδηγίας στην ισότητα στην απασχόληση, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά και επισημαίνει την ανάγκη συνδυασμού της υφιστάμενης νομοθεσίας με δράση πολιτικής και την βελτίωση της ε, συνειδητοποίησης των δικαιωμάτων με βελτίωση και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Επίσης η έκθεση τονίζει και άλλες πτυχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει το έπακρο την οδηγία σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, προωθούμε ανάλυση και έρευνα της κατάστασης στα κράτη-μέλη μέσω της ετήσια συγκριτικής έκθεσης ε, για τις διακρίσεις στην Ευρώπη που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση, την έκθεση για τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, την έκθεση για τις ε, διακρίσεις εις βάρος αναπήρων και το πώς εφαρμόζεται η οδηγία στην κρατημέλη και τέταρτον μία ε, έκθεση για τις πολλαπλές διακρίσεις, για την ισότητα των φύλων και την απαγόρευση των διακρίσεων. Και επίσης ε, θέλουμε να συγκεντρώνουμε ακριβείς και ποιοτικέ ε, πληροφορίες. Βέβαια, όλες αυτές οι εκθέσεις από μόνες τους δεν αποτελούν λύση, αλλά η ε, καλύτερη ανάλυση των τρόπων διάκρισης θα μας βοηθήσει να χαράξουμε τις κατάλληλες πολιτικές και να πετύχουμε την εφαρμογή τους. Επίσης, η, ομάδα υψηλού επίπεδου για την ισότητα και την πάταξη των, πρακτικό των διακρίσεων βελτιώνει ε, την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιση των πρακτικών. Επίσης, με την ενίσχυση της πρόσβασης στη, δικαιοσύνη, ε, ε, ενισχύουμε τους εθνικούς φορείς, μάλιστα οργανώνουμε σεμινάριο όπως αυτό το 2015 για τα θεμελιώδη δικαιώματα που επικεντρώνεται στην ανοχή, στο σεβασμό και στην καταπολέμηση ε, του αντισημιτικού ή αντιμουσουλμανικού μίσους ή μυσαλλοδοξίας και την αποφυγή των πολλαπλών διακρίσεων. Επίσης, συνεργαζόμαστε με πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο θέμα της πάταξης των διακρίσεων, την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το EQUINET, το Δίκτυο Εθνικών Φορέων Πρόθεσης Ίσης Μεταχείρισης. Επίσης, Είχαμε την πρόταση του 2008 για την οδηγία της ε, ίσης μεταχείρισης. Έτσι, επεκτείνουμε την απαγόρευση της διάκρισης λόγω θρησκείας υπευθύσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού και σε κλάδους που δεν καλύπτονταν μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, το θέμα της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών ε, εκτιμάτων, πρόσβαση στην παιδεία και παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, ενισχύουμε την προστασία ε, και από διακρίσεις λόγω ε, φύλου και ε, φιλής Γιατί αυτή το τομείς δεν καλύπτονται προηγουμένω από την οδηγία. Θεωρώ ότι η νέα πρόταση θα υιοθετηθεί σχετικά σύντομα από το Συμβούλιο. Επίσης, σημειώσαμε πρόοδο και στα θέματα της προτινόμενης οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και η πρόοδο αυτή είναι ορατή και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Η προσβασιμότητα θα είναι καταλήτη για την ίση και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και των ατόμων με ειδικέ ανάγκε ή με αναπηρίε. Επίση, θα ήθελα να ξέρω το έντονο έργο που γίνεται σε σχέση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίε και την ε, επικείμενη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για, τη, για τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης, το 2015 προτείναμε ένα πλήρη κατάλογο δράσεων για να αποφύγουμε τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ. Και ας μην ξεχνούμε και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ερμηνεύει το εύρος ε, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαίου κατά των διακρίσεων. Περιμένουμε σημαντικές αποφάσεις για δύο ε, κρεμείς για δύο κρεμείς υποθέσεις για μουσουλμάνες και το δικαίωμά τους να φέρουν τη μαντήλα στο χώρο εργασίας. Επίσης, ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας ε, θα γίνει δυνατή μόνο με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, γιατί οι δημόσιες αρχές βοηθούν στην αύξηση των εφοδίων των προσόντων ε, των εργαζομένων, αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν να δεσμευτούν για υπέρ της διαφορετικότητας και χάρη σε αυτήν να υποφεληθούν από διευρυμένη καινοτομία, παραγωγικότητα και επιδόσεις. Τα συνδικάτα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει αλλά και τα πανεπιστήμια μπορούν να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους και να μεταδώσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, τις διαφορετικότητες και τις αποφύγει των διακρίσεων. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων η κυρία Στίβενς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από αυτή την Επιτροπή, την έκθεση με σχόλια προκύπτει 60 χρόνια μετά την ε, έγκριση της ε, σχετικής ε, συνθήκης υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού Λιγότερο από το 50% των ατόμων με αναπηρία έχει ε, μια θέση εργασίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση από όλους τους τομείς με μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ιδιαίτερα το ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης, κάτι το οποίο συχνά δεν συμβαίνει. Παραδείγματο χάρη, εργαζόμενοι με αναπηρία συχνά αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια και διοικητικά, ενώ βεβαίως οι εργαζόμενοι χωρίς αναπηρία δεν έχουν τέτοια ζητήματα, κατά το οποίο είναι απαράδεκτο. Τέλος, χαίρομαι για το ότι η έκθεση παραπέμπει στην, στην ε, σχετική συνθήκη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Την μοναδική παγκόσμια τέτοια συνθήκη, την οποία έχει κυρώσει η Ένωση. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Βέμπερ, την εισηγήτριά μας για την έκθεσή της. Συμφωνώ μαζί της ότι η διάκριση στο χώρο εργασίας είναι όντως πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση στον τομέα αυτό. Συνέταξε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών ε, για το θέμα της ισότητας στην απασχόληση. Στην γνωμοδότησή μου επισημαίνω το πρόβλημα των πολλαπλών διακρίσεων και μερικές φορές και των έμεσων διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Έτσι έρχονται σε δυσμενή θέση λόγω της μητρότητας, για παράδειγμα. Επίσης, οι γυναίκες αναλαμβάνουν κυρίως τις φροντίδες του σπιτιού. Ε, θα πρέπει το έργο τους να αναγνωρίζεται και να μπορούν να συνεχίσουν ε, την εργασία τους. Να μην ε, έρχονται σε δυσμενή θέση λόγω της μητρότητας ή της φροντίδας άλλων προσώπων. Επίσης, θα πρέπει ε, η Επιτροπή να κάνει νέες προτάσεις. Είναι βέβαια δύσκολο να προβούμε σε εναρμόνιση για θέματα ηθικής ιδεοντολογίας ή να επικρίνουμε τα κράτη-μέλη επειδή απαγορεύουν ε, την ε, χρήση θρησκευτικών συμβόλων στον χώρο εργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη και να αφήσουμε σε αυτά τη διακριτική ευχαίρεια να ρυθμίσουν τέτοια θέματα. Εμεί θα πρέπει να προωθούμε την ισότητα στην απασχόληση. Αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εφαρμόσουμε.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 επεκτείνει την ε, προστασία κατά των ε, διακρίσεων. Όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο λοιπόν, εντός του οποίου πλαισίου μπορεί κανείς να καταπολεμήσει τη διάκριση που γίνεται βάσει ε, πίστης, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας κλπ. Και στόχος είναι στις χώρες μας να εφαρμόζουμε μια ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων χωρίς ε, να υπονομεύεται όμως και ο ρόλος των χωρών. Πρέπει να έχουμε τις εγγυήσει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μοιράζονται αυτή την πρακτική και άλλες χώρες και να βασιστούν στην δημιουργηθή σε εμπειρία ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν κόσμο που είναι πιο ανεκτικός ε, και να μειωθούν οι διακρίσεις. Κάζα, έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Τσάνι.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 δουλειά να κάνουν. Κυρίως ε, κάποια κράτη-μέλη που έχουν ε, μείνει λίγο πίσω. Έχετε όμως την αίσθηση ότι τα μέτρα τώρα στο επίπεδο κρατών μελών η Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα καταστήσουν δυνατόν τα παιδιά με αναπηρία να... για την απάντηση. Naturalment, sur President, fil li. Βεβαίως, ε, Πρόεδρε, μίλησα υπέρ της μειώσεως των διακρίσεων. Δεν είμαστε τέλειοι, πολλά πρέπει να γίνουν. Βέβαια, αρκετές χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν διακρίσεις θα πρέπει να κινηθούν. Να δούμε πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες όπως προανέφερα, τόσο ώστε όλοι μαζί να μπορούμε να εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα της διάκρισης από όλες τις χώρες. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Μπλίνσκεβισιούτε. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai dėkoju pranešėjai Renatai Weber už gerą pranešimą ir už mūsų bendradarbiavimą. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, έκθεση αυτή και τη συζήτηση. Η έκθεση αυτή επηρεάζει την καθημερινή ζωή ε, των πάντων ε, ανθρώπων με αναπηρία, ανδρών, γυναικών είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη και την αύξηση, στην, την αύξηση των ορίων ηλικίας δεξιοδότησης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων και καθώς βεβαίως ανεβαίνει η ηλικία συνταξιοδότηση πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ευκαιρίες για αυτούς τους εργαζόμενους για να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω από τα μελη να προστατεύουν τους πιο ηλικιωμένους από τις άδικες απολύσεις ε, λόγω ηλικίας γιατί γίνονται εύκολος ε, στόχος. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι βεβαίως η πιο ευπαθής ομάδα της κοινωνίας μας, τα άτομα με αναπηρία. Πολλά κρατημέλη παραβιάζουν την ε, οδηγία καθώς δεν έχουν προσαρμόσει το περιβάλλον εργασίας στις ανάγκες των αναπήρων και δεν έχουν διασφαλίσει ε, τις ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη-μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία και να προσαρμόσουν το χώρο εργασίας στις ανάγκες των αναπήρων. Τρίτον, είναι σημαντικό να δούμε το θέμα της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας που μπορεί να σχετίζεται με το φίλο την ηλικία, θρησκεία ή τα πιστεύω. Αυτό βλάπτει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται οι εργαζόμενοι σε τέτοιο περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει διάδοση των πληροφοριών και ενημέρωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για την ευθύνη των εργοδοτών. Οι περισσότεροι πολίτες μας δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα που τους δίνει αυτή η οδηγία. Και μεταρρυθμιστών το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Τρεμπέσιος. E Σας ευχαριστώ. Η ομάδα μας υποστηρίζει μέτρα κατά της διακριτικής μεταχείρισης στον χώρο εργασίας, όμως επίσης θεωρούν πως η οικονομία μας δεν μπορεί να επιβαρύνεται υπερβολικά με ρυθμίσεις οι οποίες τελικά κοστίζουν θέσεις εργασίας. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενη για το ότι η έκθεση αναφέρει και το θέμα της καλύτερης νομοθεσίας. Όπως σε κάθε νομοθετική έκθεση πρέπει να προσέξουμε να επιτευχθούν οι στέοχοι χωρίς κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν στις προθέσεις μας. Βεβαίω το Συμβούλιο Υπουργών δεν κατέληξε σε έναν συμβασμό, οπότε θα πρέπει να επανεπεξεργαστούμε τη σχετική οδηγία. Τέλος, δύο παρατηρήσεις. Εμείς δεν θα στηρίξουμε την κοινωνική ρήτρα στις δημόσιες προμήθειες, όπως και την ε, κατεπίγουσα εισαγωγή μιας διάταξης για την αδιαμετρότητα. Αυτό είναι εθνική υπόθεση. Των φιλελευθέρων και δημοκρατών το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Χάρκη. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Η Ρενάτα Βέμπερ ε, παρήχε πλήρη, ε, μια παρήχη έκθεση όσον αφορά τις προκλήσεις που έχουμε όσον αφορά την ισότητα στην απασχόληση. Κάποια από τα προβλήματα και τις προκλήσεις ήδη αναφέρθηκαν από την Επίτροπο, την κυρία Τάισεν. προηγουμένω η έκθεση ασχολείται με βασικά θέματα όπως αναπηρία, ηλικία, θρησκεία, ε, πίστη, σεξουαλικός προσανατολισμός, αλλά βλέπει και οριζόντιες πτυχές που σχετίζονται με αυτά. Κάποια θέματα είναι πιο εύκολα και προσμετρώνται και πιο εύκολα, όπως η παροχή λογικής στέγασης για ανθρώπους με αναπηρία, η χρήση σχεδιασμού ειδικού σε διάφορες δημόσιους χώρους, οι κοινωνικές ρήτρες, οι διαδικασίες κρατικών προμηθειών, να δούμε ποια είναι τα ενότητα, τα όρια ηλικία για κάποιε τη απασχόληση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση ε, διαφόρων ρυθμίσεων όσον αφορά γονικά δικαιώματα, γάμους κλπ. Κάποια θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ευαίσθητα. Άρα έχουν σοβαρό αντιχτύπο εθνικό επίπεδο. Καμιά φορά λόγω πολιτισμού, ιστορίας και πιο προσφάτων γεγονότων. Και αυτό που έχω να πω σε αυτό είναι ότι όταν δικαιολογεί κανείς τη διάκριση στον τομέα της απασχόλησης σε αυτά τα θέματα, τότε ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για 1,5 λεπτό η κυρία Κάρη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την κυρία Βέμπερ, για την πολύ αξιόλογη της έκθεση. Πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα μας αφορά όλους. Το θέμα της ε, πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους, άσχετα με την θρησκεία, γενετήσιο προσανατολισμό, εθνοτική καταγωγή και ούτω καθεξής. Οι ίσεις, ε, οι ευκαιρίες θα πρέπει να αποτελέσουν καθήκον μας, γιατί δυστυχώς πολλοί συμπολίτε μας βιώνουν διακρίσεις. Για παράδειγμα, οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην πρόσβαση ε, σε συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης και υπάρχει ακόμη και μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης ε, και κάποιες ε, μειονοτικές ομάδες ε, έχουν πρόβλημα στην ένταξη στην αγορά εργασίας και έχουν χαμηλότερους μισθούς. Για μερικούς συμπολίτες μας είναι τελείως αδύνατη η πρόσβαση στην αγορά εργασίας εξαιτίας των διακρίσεων. Θα πρέπει αυτές οι διακρίσεις να σταματήσουν. Να επιτρέψουμε επίσης τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε περισσότερες και πιο ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να πατάξουμε τις διακρίσεις. Αυτό θα ωφελήσει. Μας είναι συλλογικό το έργο και όχι ατομικό πρόβλημα. Των πρασίνων το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ζντάνοκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη Ρανάτε Βέμπερ για την έκθεσή της οι πράσινοι στηρίζουν πλήρως την έκκληση προς το Συμβούλιο να διακόψει επιτέλους αυτή την αποτελμάτωση το αδιέξοδο και να επισπεύσει την, την υιοθέτηση μιας οριζόντιας οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πάταξη των διακρίσεων. Έχουμε κάποια μέτρα κατά των διακρίσεων, αλλά δεν εφαρμόζονται δυστυχώς ομοιόμορφα από τα κράτη-μέλη. Μία τέτοια ομοιόμορφη εφαρμογή θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις. Η σχετική οδηγία δίνει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προβλέψουν κάποια θετικά μέτρα για ομάδες που υπόκεινται πολλαπλές ή διαρθρωτικές διακρίσεις. Δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται στο έπακρο η οδηγία αυτή από τα κράτη-μέλη. Επίσης, Συμφωνώ με τη σύσταση να εθετηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών για να καταπολεμηθεί η Ισλαμοφοβία και ο αντισημιτισμός. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω και τη ρωσοφοβία. Είναι ένα σχετικά νεοφανές φαινόμενο. Για την ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Τζέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τη συνάδελφο την κυρία Βέμπερ για τη δουλειά που έκανε. Η οδηγία γεννάται, γεννήθηκε εδώ και 16 χρόνια και αν δεν λάβουμε υπόψη πώς εφαρμόστηκε αυτά τα χρόνια, πιστεύω παρόλα αυτά ότι η δουλειά που έγινε είναι θεμελιώδου σημασία. Διότι κατά τη διάρκεια τη χρονική περίοδου τα διαθροτικά προβλήματα των κρατών μελών δημιούργησαν νέε ανισότητε. Έχουμε νέα τμήματα του πληθυσμού και κυρίως εντός της αγοράς εργασίας που υπόκεινται σε ανισότητες όπως είναι άνθρωποι στους οποίους επευλήθη ε, μία αύξηση του, συνταξι... του έτου συνταξιδότησης και κατά κάποιο τρόπο είναι θύματα διακρίσεως διότι δεν έχουν επαρκείς δεξιότητες να προσαρμοστούν στην αλλαγή της αγοράς εργασίας όπως και τα άτομα που είναι θύματα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης